Welcome back to Καλώς επιστρέψατε. Καλώς ορίσατε στην συνεδρίαση των συντονιστών στη συνεδρίασή μας. Καλώς ορίσατε και όσοι δεν συμμετείχατε στη συνάντηση των συντονιστών. Καλώς ορίσατε και συντονιστές. Έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα, πολλές δύσκολες ε, ε, αναφορές θα πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ας εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Δεν έχουμε να εγκρίνουμε πρακτικά. Έχω δύο παρατηρήσεις. Η διαμεσολαβήτρια θα είναι εδώ στις 11, όπου θα πρέπει να κάνουμε τις ψηφοφορίες γρήγορα. Βρίσκεται ήδη καθοδόν και αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα εργαστούμε πολύ γρήγορα γιατί έχουμε στενά περιθώρια. Οπότε θα έχουν δύο λεπτά όλοι οι συνάδελφοι για παρεμβάσεις, όχι παραπάνω. Υπό τα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Και ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα η γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Βάλτε τις κάρτες ψηφοφορία σας, ε, αν τις έχετε μαζί σας ε, και θα ξεκινήσουμε άμεσα. Okay, this is going to be a little bit complicated vote. Θα είναι λίγο περίπλοκη η ψηφοφορία προ το παρόν. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν τροπολογίε τι οποίε θα πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Και ούτω θα πράξουμε. Θα σας το πω θα φτάσουμε σε αυτές. Λοιπόν, ε, σχέδιο γνωμοδότησης τη Επιτροπής. Ζητά συγγνώμη η Πρόεδρος. Δεν είμαι άρρωστη, η γύρι είναι, αλλεργία. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε στην τροπολογία 96, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 98 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97, επίσης σε δύο τμήματα, ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, Καταπίπτει 97. Ωραία. Λοιπόν. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 105 Καταπίπτει, καταπίπτει όπως το είπατε, να αφού η άλλη εγκρίθηκε ήδη. Πάμε στην 2.50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.51. Καταπίπτει. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. And now we can close the vote. Πέρας εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω αλλά να ελέγξουμε έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται Τροπολογία 118 και 119 είναι ταυτόσιμες επί της ουσίας. Ας τις ψηφίσουμε μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 56. Περνάμε σε αυτήν. Έχετε δίκιο. Όχι, μπορούμε να ψηφίσουμε την 56 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά να ελέγξουμε ποια λέτε 132 έναρξη ψηφοφορίας για ηλεκτρονικό έλεγχο της 132 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 Καταπίπτει. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το μπλοκ 1 έχει αποσυρθεί το μπλοκ 2 επίσης και το μπλοκ 2 και το μπλοκ 3 καταπίπτουν κινούμαστε πολύ γρήγορα τροπολογία 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ Εγκρίθηκε με τη συμβιβαστική. Είναι λίγο περίεργη η λίστα αυτή. ...174 τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ καταπίπτει συγγνώμη 100 η θεωρείται ότι έχει υιοθετηθεί με τη συμβιβαστική 9. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει επίσης συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα αιτιολογική σκέψη 22α τροπολογία 68 αυτή πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά. Με ακούτε? Με παρακολουθείτε? Δεν με παρακολουθείτε. Είναι λίγο μακριά. Υπό τη συμβιβαστική 9 στο τέλος η αιτιολογική σκέψη 22α τροπολογία 68 θα πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά. Είναι τροπολογία της Ελεονόρα του Φάμπιο Μάσιμου πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά. Ζητάτε το λόγο επίσημα γιατί δεν σας ακούω όταν μιλάτε όλοι μαζί. 68 τροπολογία. Πρέπει να τη βγάλουμε από τη συμβιβαστική και να την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Μαρλένα, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 210, ε, γιατί εκεί έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Sorry about that. We need... Ζητώ συγγνώμη. Πολύ σωστά το είπε η Μαρλένε. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 210 κατά τμήματα. Για το δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε. Απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 68. Την ψηφίζουμε ξεχωριστά. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Από εκεί πάμε στην 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 προφορική τροπολογία των πρασίνων. Έχετε το κείμενο ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ έχει εγκριθεί οι 2 02 μέχρι 205 καταπίπτουν πάμε στη 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβεστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έχουμε την τροπολογία 219 που θα ήθελαν ε, οι πράσινοι να συμπεριληφθεί. Είναι προφορική τροπολογία. Μπορούμε να την ψηφίσουμε. Δεν την προσβάλλει ο εισηγητής, οπότε δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Καταπέπτει μαζί με τη συμβιβαστική 2.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.25 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 2.26 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε The Πέρας. Εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά. Κοιτάξτε, κάνετε τόσο πολύ θόρυβο. Πρέπει πραγματικά να γνωρίζω ποιος ψηφίζει. Μη μιλάτε όλοι μαζί και μιλάτε δυνατά. 227 ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ, άρτη ψηφοφορία. It has been adopted. Εγκρίνεται. 228 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 12, την τροπολογία 229, δηλαδή το δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 231 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94. Η καταπίπτη με συγχωρείτε. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ψηφίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία τη 243. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν τη 241 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 242 υπέρ. Καταπίπτει 244 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 245 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 245 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεν ψηφίζεται όμως. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 248 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές αναφορές, τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική παλήθευση για τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία. Γκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε, με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημασική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά όχι, όχι, δεν καταπίπτει. 26. Πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. ουδείς, Λέει ότι καταπίπτει στην πράξη δεν καταπίπτει. Έχει γίνει λάθος. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την 26 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές το πρώτο τμήμα, λέει πρόεδρο και εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τη 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, Αποχέ απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, η καταπίπτη μάλλον. Η 35 έχει αποσυρθεί, 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. καταπίπτη 37, αλλά ψηφίζουμε την 38. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν μπορώ να δω τελικά πώς ψηφίζετε. Έχετε κουραστεί, το καταλαβαίνω. Ψηφίζουμε πάλι την τροπολογία τη 42 ψηφίζαμε. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 47 καταπίπτει και η 48, 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 56. Στη 57 μάλλον διορθώνει η Πρόεδρος, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ. Την 65 ψηφί έχει εγκριθεί. Την 65, την 65. Βιαζονή, παρακαλώ, έχει το λόγο. Έχει γίνει λάθος μάλλον με τον κατάλογο ψηφοφορίας. Εγκρίναμε την 63. Οι επόμενες δύο πρέπει να καταπέσουν, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι, είναι συμβατές. Πρέπει να τι ψηφίσουμε, λέει πρόεδρος. Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε 65 υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο πλαίσιο της συμβαστικής αυτής τροπολογίας, στο 69, δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 79. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ υπέρ της 80 παρακαλώ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 80 όχι δεν καταπίπτει έχει γίνει λάθος εδώ στον κατάλογο ψηφοφορίας 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 καταπίπτει 85, περνάμε στο 86 σε δύο τμήματα. Α, 87 λοιπόν, Ψηφίζουμε την 87. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Πολύ ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 89. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 91 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε, στην 84, στην τροπολογία 84 λέει αν εγκριθεί πηγαίνετε στην τροπολογία 88. Πού βρίσκεται αυτή η τροπολογία 88, δεν υφίσταται τέτοια τροπολογία. Όντω δεν υφίσταται. Έχει γίνει λαθασμένη ένδειξη εδώ πέρα στον κατάλογο ψηφοφορία. Δυστυχώ ο κατάλογο αυτό ψηφοφορία βρήθη λαθών. Λοιπόν, α περάσουμε στη ηλική ψηφοφορία, λέει Πρόεδρο. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ο Ομόφωνα εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Να σας εξηγήσω τώρα τι έγινε με την ψηφοφορία αυτή. Λόγω του ότι είχαμε νέα μέλη στο προσωπικό μας, δηλαδή από ανθρώπινο σφάλμα ο κατάλογος αυτός δεν ήταν καλός. Υπήρχε σήμερα μελέτη συνδελεχέστατα τη λίστα ψηφοφορία. Σήμερα δεν θα επαναληφθεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Πρόκειται για προφορική ερώτηση Okay, so the, the... Λοιπόν, προφορική ερώτηση για απάντηση από την Κομισιόν σε σχέση με την αντιμετώπιση των αναφορών για την αντιμετώπιση της επισφάλειας και καταρχής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is now. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Επόμενη ψηφοφορία. Αντιμετώπιση των αναφορών σχετικά με την αντιμετώπιση επισφάλειας και έτσι καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Τζουντ, ναι, μια ενημέρωση. Θέλουμε να αποσύρουμε δύο τροπολογίες, ε, ε, την 46 ε, και την 50. Το ξέρει η γραμματεία, απλά για να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Πολύ καλά, λέει πρόεδρο. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Μετά έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες που έχουν αποσυρθεί, Αρκετέ, αρκετέ. Τροπολογία 10. Από κοινού δεν είναι τη ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Να ελέγξουμε θέλετε την 10, να την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τη 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 έχει αποσυρθεί και η 21. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία α. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία Β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Σ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 35-39 έχουν αποσυρθεί. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 41 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε 43 απλά και μόνο γιατί τα χέρια όχι γιατί δεν είναι σαφές υπεράριθμοι από το ΕΛΚ ένας παραπάνω τώρα εντάξει εγκρίθηκε οι 44 και 45 ταυτόσιμες ψηφίζουμε από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 46 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική ή ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 αποσύρθηκε. Άρα ψηφίζουμε την 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 53. Πέραση ψηφοφορίας. πράγματι απορρίφθηκε. Πηγαίνουμε στην 54 ψήφι πέρα κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Όχι. Θα την ελέγξουμε. 58. Απορρίφθηκε. 59 υπέρ. Υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, ελέγχουμε την 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε 63. 64 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 67, 68, συγγνώμη, 67 και 70 έχουν αποσυρθεί. Ψηφίζουμε την 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 72. Δεν έχουμε τμήματική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της 72. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει για την 73. Δεν είναι τμήματική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε όλη την τροπολογία από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 θέλετε να ελέγξουμε την 75 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε που πάω τώρα 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81, 2, 3, 4, 5 έχουν αποσυρθεί πηγαίνουμε σε συμβαστική H ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πηγαίνουμε στην 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Σφάλμα μου. Μάλλον δεν έχω ξυπνήσει καλά ακόμα. Είπα λάθος ε, αποτέλεσμα. Άι, συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, ελέγχουμε την 98. Αγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Πηγαίνουμε στην 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103-104 ταυτόσημες. ψήφισαν από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 105 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν ε, βλέπω τα χέρια, να ελέγξουμε λοιπόν και την 105. Απορρίφθηκε. Πηγαίνουμε στην 106. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109. Ψήφι υπέρ. Όχι. Καταπίπτει.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 Πηγαίνουμε στην 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και τώρα, που πάμε. Exactly. Now, uh, item A. Περνάμε στο σημείο 8, το οποίο θα έπρεπε να το δούμε τώρα, αλλά ε, πρέπει να περάσουμε πρώτα στη διαμεσολαβήτρια γιατί βιάζεται οπότε θα αναβάλουμε την διερευνητική επισκέψη θα την δούμε το απόγευμα οπότε ας καλέσουμε την Έμιλη Οράιλη να πάρει το λόγο colleagues, please. Αγαπητοί συναδελφοί, παρακαλώ καθίστε. Δεν θα έλεγα να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας. Αλλά καθίστε και όσοι είναι να φύγετε από την αίθουσα παρακαλώ φύγετε. Αποχωρήστε ησύχω με λίγο σεβασμό στις εργασίες μας. Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω σήμερα το πρωί την Έμιλη Ωραίλη, ε, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, να μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του 2017 στην Επιτροπή μας χωρίς άλλη καθυστέρηση. Έχετε το λόγο. Uh, thank um, Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να βρίσκομαι εδώ σήμερα και που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μας για το 2017. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, εξαιρετικά την Επιτροπή σας μας έχετε προσφέρει τεράστια υποστήριξη στην υπηρεσία μου πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό για μας το να λαμβάνουμε τόσο μεγάλη ε, διαρκή υποστήριξη και σε επίπεδο γραφείου και σε ατομικό, σε προσωπικό επίπεδο με τους ευρωβουλευτές που συναντούμε σε άλλο πλαίσια. Σας ευχαριστούμε λοιπόν να ξεκινήσω. Πέρυσι διεκπαιρεώσαμε λίγες παραπάνω από 2.000 καταγγελίες. Ανοίξαμε πάνω από 400 έρευνες βάση καταγγελιών και 14 έρευνες ε, ιδίας πρωτοβουλίας. Ιδίας πρωτοβουλίας γιατί πολύ συχνά έχουν να κάνουν με ζητήματα υψηλού ε, ενδιαφέροντος ε, με μεγάλη προβολή στον τύπο. Ε, πάνω από το 75% των καταγγελιών ε, των ερευνών που κάνουμε είναι ατομικές καταγγελίε από πολίτες, από βουλευτές, από ΜΚΟ, από την κοινωνία των πολιτών κτλ. από πού προέρχονται οι περισσότερες καταγγελίε δεν έχει αλλάξει η κατάσταση από τα προηγούμενα έτη. Ο υψηλότερος αριθμός έρχεται από την Ισπανία λόγω του, του πληθυσμού της χώρας αλλά και λόγω του αναπτυγμένου συστήματος ε, ε, διαμεσολαβητής ε, τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Είναι συνηθισμένοι οι Ισπανοί σε αυτό το θεσμό του διαμεσολαβητή. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε τόσο πολλέ καταγγελίε από και Η Γερμανία και η Πολωνία πάλι, επίση από του πρώτου, λόγω των μεγάλων πληθυσμών του. Και πολλέ φυσικά καταγγελίε από το Βέλγιο για του σαφεί λόγους ότι εδώ βρίσκονται θεσμικά όργανα, πολλές ΜΚΟ, πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών βρίσκονται εδώ στο Βέλγιο, γι' αυτό λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες και από το Βέλγιο. Στην επόμενη διαφάνεια επίσης θα δείτε κάτι εκεί, οι περισσότερες καταγγελίες είναι κατά της Κομισιόν, όχι για την κακή της διοίκηση αλλά γιατί παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στις ζωές όλων μας. Γι' αυτό οι περισσότερες καταγγελίες τρέφονται κατά αυτόν. Η έψω από ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν δουλειά εδώ στα θεσμικά όργανα και θεωρούν ότι αδικήθηκαν κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι για τον πολιτικό του ρόλο αλλά για το διοικητικό του ρόλο ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, ε, η Όλαφ ε, λαμβάνουν καταγγελίες επίσης λόγω τρόπου διεξαγωγής ερευνών και άλλα, άλλοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε αυτό που θεωρώ εγώ ένα από τα πιο επιτυχημένα μας, μια από τις πιο επιτυχείς μας υποθέσεις πέρυσι Πρόκειται μια καταγγελία Αυστριακού πολίτη, ο οποίος εργαζόταν ως εκπαιδευόμενος σε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ασία, χωρίς αμοιβή, όπως όλοι οι εκπαιδευόμενοι, όχι απλά χωρίς αμοιβή, αλλά χωρίς ε, καν έξοδα ταξιδιού, ε, διαμονής και διατροφής. Τίποτα. Θεώρησε ότι ήταν άδικο, ότι αποτελούσε διακριτική μεταχείριση και εμεί θεωρούσαμε ότι αυτό ε, απορρέει από τι συνθήκε ω απέτηση να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση προ του νέου αυτού τους ανθρώπους οι οποίοι καταφέρνουν επιτέλου να επιτύχουν μια ε, τέτοια εκπαίδευση για να κάνουν μια τέτοια εκπαίδευση χωρίς αμοιβή είναι γιατί οι οικογένειές τους έχουν χρήματα και είναι κρίμα γιατί άλλοι άνθρωποι επίσης ε, ε, ικανοί δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν τέτοια εκπαίδευση γιατί δεν έχουν υποστηριχθεί από τις οικογένειές τους οπότε ζητήσαμε επανεξέταση αυτή τη υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και η Επίτροπος κ. Μουγκερίνη απάντησε πολύ θετικά. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι το Συμβούλιο συμφώνησε προπολογισμό λίγο παραπάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ και το Κοινοβούλιο επίση. Και έτσι οι εκπαιδευόμενοι στο μέλλον θα αμείβονται. Ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό από το Κοινοβουλίο και το Συμβούλιο άλλες ε, καταγγελίες με ε, καλή έκβαση. Ε, μια από τις κλασικές καταγγελίες που λαμβάνουμε είναι προσπάθεια ανάκτησης χρημάτων της Κομισιόν από μια βελγική ΜΚΟ λόγω προβλημάτων διεξαγωγής των εργασιών παρότι παραδόθηκε επιτυχώς το έργο. Μετά από την έρευνά μας το ποσό που ζήτησε η Κομισιόν μειώθηκε κατά περίπου 37.000 μεγάλη ανακούφιση για την ΜΚΟ μια άλλη καταγγελία κατά του ΕΦΣΑ μια γαλλική ένωση διαμαρτυρήθηκε για μια αξιολόγηση ε, γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού η πρόταση έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων την ΕΦΣΑ έγιναν δεκτές και οι συστάσεις βελτίωση για το μέλλον ε, όσον αφορά όλε αυτέ τι άδειε ώστε ο κόσμο να είναι βεβαίω ότι η δουλειά γίνεται αποτελεσματικά σωστά και σωστά. Και εδώ βλέπετε μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε πέρυσι πιλωτικά. Είναι κάτι πρόσφατο. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος ε, ενοχλήθηκε από τον πολύ χρόνο που χρειάστηκε ε, για να έχουμε καταγγελίες σε σχέση με την άρνηση ε, παροχής ε, πληροφοριών εγγράφων από την Κομισιόν και από άλλα θεσμικά όργανα. Το κοιτάξαμε και αντιληφθήκαμε ότι υπήρχε ένα βήμα στη διαδικασία το οποίο μπορούσαμε να βγάλουμε. Για να σας το εξηγήσω απλά, αφού λαμβάνουμε την καταγγελία, ε, ζητάμε στην Κομισιόν, ας πούμε, αν ζητήθηκε από την Κομισιόν να απαντήσει, παρότι θα ήταν κατανοητή η απάντηση που δόθηκε στον Ατούντα, ε, καθυστερούσε η Κομισιόν ε, τη διαδικασία. Από σε συνεργασία με την Κομισιόν αποφασίσαμε να βγάλουμε αυτό το βήμα και τώρα η διαδικασία είναι πιο γρήγορη όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα. σκοπό μου είναι να λαμβάνετε απόφαση εντός 40 ε, εργάσιμων ημερών. Και αυτό το ζήτημα σας είναι επίσης γνωστό γιατί ακούγεται εδώ και χρόνια. Με μεγάλη μου χαρά η Κομισιόν έλαβε υπόψη κάποιες από τις συστάσεις μου σε σχέση με τη βελτίωση του κώδικα διοντολογίας που τρέχει αυτή τη στιγμή ώστε το cooling off period, η περίοδος αναμονής να παρατείνεται ε, τόσο για τους επιτρόπους όσο και για τον πρόεδρο της Κομισιόν. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, όχι αρκετές πιστεύω, αλλά πολλές από αυτές τις αλλαγές ε, θα είναι εξελικτικές όχι επαναστατικές. Οπότε χαίρομαι που η Κομισιόν έλαβε υπόψη πολλά από αυτά που προτείναμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Έκτοτε έχω ε, στραφεί στην Κομισιόν και τους έχω γράψει ε, σε σχέση με καταγγελίες που έχουμε λάβει όσον αφορά τον τέος πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόσο, ανοίξαμε μια έρευνα, κάναμε συστάσεις και τώρα εξετάζουμε την απάντηση της Κομισιόν, η οποία ήταν αρνητική κατά κάποιους τρόπους. Οπότε εξακολουθούμε τη μελέτη. Γενικά όμως ε, έχουν παρατευθεί και αλλαγές και βελτίωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Κάτι που πιστεύω είναι σημαντικό για τους πολίτες ε, και για άλλους φορείς. Έχουμε λάβει όπως γνωρίζετε δύο καταγγελίες από δύο αντιπροσωπείες ε, ευρωβουλευτών για, την πρόσφατο, για τον πρόσφατο διορισμό του Μάρκου Σέλμα, ιεροσγενικού Γραμματέία της Κομισιόν Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ε, έχει μελετήσει εκτενώς το θέμα αυτό, το έχουμε παρακολουθήσει στενά. Όπως έχω ξαναπεί στην Επιτροπή αυτή, δεν θέλουμε να, να επαναλαμβάνουμε τη δουλειά άλλων, ε, ειδικά όταν είναι επιτυχής, διότι αυτό αποτελεί σπατάλη πόρων. Αλλά έχουμε υποβάλει κάποια ερωτήματα στον Πρόεδρο Γιούνκερ και ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχει η Κομισιόν στα χέρια της και ο έλεγχος αυτός θα θέλαμε να λάβει χώρα μέχρι τις 8 Ιουνίου. Θα σας στηρίσουμε ενήμερος λοιπόν για το θέμα αυτό. Και εδώ έχουμε μια άλλη καταγγελία που βρίσκεται αρκετό καιρό στις υπηρεσίες μας σχετίζεται με την ε, ιδιότητα μέλους του Πρόεδρου της ε, Κεντρικής Τραπεζάς του κ. Μάριο Ντράγκη ε, Group of 30 ε, μια ένωση ε, τέος και σημερινών τραπεζιτών, ε, προέδρων κεντρικών τραπεζών, η καταγγελία ισχυρίζεται ότι, το, ότι ο κύριος Ντράγκη είναι μέλος αυτής της ομάδας είναι κάτι διαφανές και ασύμβατο με την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ξέρετε έχει τεράστια αυτονομία λόγω του ρόλου της. Ε, ε, υποτίθεται ότι αποφεύγεται οποιαδήποτε παρέμβαση στι εργασίες τη, Οπότε η σύσταση που έκανε ήταν ο κύριο Ντράγκη να παρατηθεί σε κάθε περίπτωση και να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Οκτώβριο του χρόνου ότι έχει αναστείλει την ιδιότητα του ως μέλους της ομάδας των 30. Αναμένοντα την ε, συνταξιοδότησή του, την αποσύρσή του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απάντησε με μια εκτενή απάντηση, αλλά μα είπε ότι η ιδιότητα μέλου στην ομάδα των 30 του κ. Ντράγκη δεν είναι ασύμβατη με τη θέση του ω Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμεί εξετάζουμε την απάντηση και την επιχειρηματολογία, τα εξετάζουμε όλα αυτά για να δώσουμε μια τελική απάντηση, μια τελική απόφαση μέσα στι επόμενε εβδομάδε για την υπόθεση αυτή. στρατηγικές μας εργασίες το 2017 ανοίξαμε τέσσερις στρατηγικές έρευνες ε, την λογοδοσία του Συμβουλίου ε, τι γίνεται με τέος προσωπικό της Κομισιόν που βρίσκει δουλειά, οκτώ στρατηγικές πρωτοβουλίες ε, με το Συμβούλιο για τη διαφάνεια του Λόμπινγκ και τη διαφάνεια του Brexit, τέσσερις στρατηγικές έρευνες για τη διαφάνεια των ομάδων εμπειρογνωμόνων και έχουμε και έξι στρατηγικές πρωτοβουλίες. Μία που σχετίζεται με τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να δούμε λίγο τους ειδικού ε, συμβούλους και τις έρευνες ε, που γίνονται σχετικά με αυτού. Ο ε, σκοπό είναι να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό είναι υπέρ των συμφερόντων όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των ειδικών συμβουλών των ίδιων, γιατί πολύ συχνά παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και δεν θέλουν κατά λάθο να βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις όπου γίνονται, υπάρχουν ισχυρισμοί για σύγκρουση συμφωνών. Έχω κάνει 10 προτάσεις εγώ στην Κομισιόν και έχουν πραγματοποιηθεί περαιτέρω βελτιώσεις σε σχέση με ε, την ε, αντιμετώπιση αυτών των συγκρούσεων συμφερόντων. Το επόμενο διαφάνεια, δικαιώματα των πολιτών και διαπραγματεύσεις για τον Brexit. Σίγουρα σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών το ζήτημα αυτό είναι... Έχει απασχολήσει το Κοινοβούλιο πολύ. Ε, λάβαμε σωστές απαντήσεις από το Συμβούλιο και την Κομισιόν σε θέματα διαφάνειας και επίσης έχουμε γράψει στον πρόεδρο Γιούνκερ ε, όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ώστε να βλέπει ο κόσμος ποιος προσπαθεί εύλογα να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ε, φαντάζομαι ότι οι πραγματικές εργασίες θα καταστούν απαραίτητε ε, όταν θα ξεκινήσουν οι εμπορικές συνομιλίες για τη μελλοντική εμπορική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η δουλειά αυτή λοιπόν τρέχει ακόμα. Μέχρι στιγμή έχει σημειώσει επιτυχία. Όπως ξέρετε η παρενόχληση έχει υπάρξει ένα παγκόσμιο πλέον θέμα. Σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς και όλους τους θεσμούς. Ε, με κάποιο τρόπο κάποιος έχει ασχοληθεί με αυτό. Ουσιαστικά δεν λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες γι' αυτό. Και σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό αυτή τη στιγμή να κάνουμε ε, μια άσκηση εγχειρήματο ε, έρευνας για να δούμε τι κάνουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να ασχοληθούν με το ζήτημα. Στον χώρο εργασία αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε πληροφορίε για τι πολιτικέ καταπολέμηση τη παρενόχληση και των σχετικών πρακτικών σε ολόκληρε τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δούμε έτσι τι κάνουν όλοι. Θα μαζέψουμε κάποιε ιδέε για να δούμε τι αποτελεί βέλτιστη πρακτική, ελπίζοντα να λάβουμε απαντήσει ε, για αυτό το θέμα μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα. Η επόμενη μας έρευνα είναι η πιο σημαντική απόψη δημοσίου ενδιαφέροντος. Την ξεκινήσαμε πέρυσι και συνεχίζεται. Αφορά τη λογοδοσία του Συμβουλίου. Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω σε αυτή την αίθουσα. Δύο βασικές συστάσεις έχουμε κάνει. Η μία είναι ότι όταν οι προπαρασκευαστικές ε, οι ομάδες, οι εργασίας ε, συζητούν ε, προτινόμενη νομοθεσία σε πρώιμο στάδιο, οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου θα πρέπει να καταγράφουν τις θέσεις των κρατών μελών. Λέμε καταγράφουν, όχι δημοσιοποιούν, όχι να τις δημοσιοποιούν σε τόσο πρώιμο στάδιο, αλλά τουλάχιστον να τις καταγράφουν γιατί εξετάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων εργασίας. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά το τι καταγράφεται και το τι δεν καταγράφεται. Και παρότι το δικαστήριο αποφάσισε το 2012 ότι δεν ε, υπάρχει κάτι που να εμποδίζει υπό την 1999 τη δημοσιοποίηση των, των θέσεων των κρατών μελών, τα κρατημέλη θεωρούν ότι αν δεν καταγράφονται οι θέσεις τους δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Μερικές φορές ο κόσμος θεωρεί ότι έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ε, δηλαδή σε αρχεία, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα αρχεία, δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Η δεύτερη σύσταση αφορούσε την ευρεία χρήση της χρήση της φραγίδας ε, περιορισμένης χρήσης, ε, απογορεύεται τη δημοσιοποίηση σε διάφορα έγγραφα και όταν ε, γίνεται αίτηση πρόσβαση σε τέτοια εγγραφά η μεγάλη πλειοψηφία τους 84 νομίζω τις 100 αυτών των ε, εγγράφων ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό τον 1999, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η σφραγίδα χρησιμοποιείται υπερβολικά και το δικαστήριο το έχει πει ξανά και ξανά. Κάθε έγγραφο πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί βάσει του περιεχομένου του. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο λοιπόν να απαντήσει μέχρι τις 9 Μαΐου ζήτησαν παράταση. Τους είπαμε ήδη ότι δεν θα τους χορηγήσουμε παράταση αφού έχουμε και εμείς χρονικούς περιορισμούς και αφού πρόκειται για ένα ζήτημα ε, υψηλού δημοσίου ενδιαφέροντος. Γι' αυτό θα ε, συντάξουμε τώρα μια ειδική έκθεση προς το Κοινοβούλιο που θα ζητήσουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Κάτι τώρα πιο ευχάριστο. Αυτή ήταν μια από τις πιο ευχάριστες εκδηλώσεις που είχαμε πέρυσι όταν καλέσαμε για πρώτη φορά όλους τους οργανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας παρουσιάσουν αυτό που θεωρούσαν αυτοί το καλύτερο του επίτευγμα σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Ε, λάβαμε πάρα πολλές υποψηφιότητες, πάνω από 90, σχεδόν 100. Ήταν μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Ε, ο κόσμος χάρηκε πολύ που αναγνωρίστηκε η δουλειά του και οι συνάδελφοι για πρώτη φορά ανακάλυψαν τι κάνουν οι άλλοι. Ε, ειδικότερα σε κάποιου οργανισμού που δεν έχουν τόση προβολή, δεν βρίσκονται στι Βρυξέλλε, δεν βρίσκονται στο Στρασβούργο ή στο Λουξεμβούργο και δεν του βλέπει κανεί ε, του χρόνου. Θα το επαναλάβουμε το βραβείο. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο στου ανθρώπου ε, να προετοιμάσουν τα έργα του και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερε υποψηφιότητε. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ και ξανά που μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ για την πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξή σας. Is... ευχαριστώ θερμά. Δεν συνηθίζεται το χειροκρότημα, το αξίζεται όμως. Πραγματικά με υποδειγματικό τρόπο δείξατε πως εσείς προσωπικά αλλά και ο φορέας σας είναι ένας φορέας επιφυλακής ε, και θεματοφύλακας ε, της εφαρμογή. Ε. Ξέρω ότι δεν μπορείτε και εσείς να παραμείνετε πολύ και εμεί είμαστε πιεσμένοι. Θα περιορίσω λοιπόν το χρονογόρευση σε 1,5 λεπτό δυστυχώς. Η Μάργκριτ όμως έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. We are very happy the Greens Είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι ως πράσινοι που πλέον ασχολείστε με τη συμπεριφορά του Συμβουλίου γιατί έχει ακόμη την οτροπία το Συμβούλιο ότι είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός και όχι ένας ενωσιακός οργανισμός. Ε, επομένως συμπεριφέρεται ως διακυβερνητικός οργανισμός. Πολλά δε ε, κυβερνητικά ε, κλιμάκια, η υπουργεία, η γραφεία δεν έχουν καταλάβει ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο συναποφασίζουμε. Πρέπει λοιπόν αυτό να το τονίσετε και θα πρέπει να προσαρμοστεί το Συμβούλιο στη συνήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμπεριληφθεί ο κοινοβουλευτικό έλεγχο, η διαφάνεια, η συμμετοχή του λαού, ώστε και τα εθνικά κοινοβούλια, ο εθνικό τύπο να μπορούν να παρακολουθούν το έργο τη κυβέρνηση τη χώρα του. Πάρα πολύ εύκολο να λέει μια κυβέρνηση. Αυτοί εκεί φταίνε αυτά τα τέρατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το τέρας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίει για όλα. Εμείς θέλουμε να προσθέσουμε και επίσης ε, παραπάνω πόρους σε εσά για να μπορέσετε να συνεχίσετε το καλό έργο. Δεν έχω κάποιον άλλο. Α, έχω την Πεατρίς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα. Καλώς ήλθατε εκ νέου κυρία Ράιλι. Πάρα πολύ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εξ ονόματος και του Χαβιέρ Νάρτε αλλά και προσωπικά εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της έκθεσης που ε, έχετε καταρτήσει. Την ε, ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως πάντα βλέπουμε ότι πρόσβαση των εγγράφων ε, και ο απολογισμός του έργου η παρουσία των διαφόρων ομάδων εργασία ε, και η διαφάνεια ενδιαφέρουν ε, το θεσμό του διαμεσολαβητή. Θέλω επίσης να τονίσω τη σημαντική συνεισφορά σας στη βελτίωση ε, της δημοκρατίας και σε ό,τι αφορά τις έρευνες και τις συστάσεις ε, ε, το έργο σας βλέπουμε ότι δίνει αποτελέσματα και οδηγεί σε μετα... μεγάλες αλλαγές. Πολύ σημαντικός ο ρόλος λοιπόν ε, του θεσμού σας και σημαντικός και ο ρόλος για την Επιτροπή ΠΕΤΗ. Θα υπάρχει στήριξη μας και στο μέλλον και ελπίζω να συνεχίσετε και εσείς το ποιοτικό έργο σας που μας βοηθά πολύ καλύτερα να κατανοήσουμε τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών.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 Ο Πέτερ Γιάρ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να ευχαριστήσω και την διαμεσολαβήτρια που πολύ σωστά είπε ε, ότι έχετε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή ε, ε, Αναφορών μας. Ευχαριστήσατε και σας ανταποδίδω τις ευχαριστίες γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το στόχο που αναφέρατε, θέλετε να έχετε μέσα σε 40 ημέρες μια απόφαση. Μακάρι και εμείς να φτάσουμε σε μια τέτοια καλή ε, απόδοση. Χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο μέχρι στιγμής για να ε, κρίνουμε μια αναφορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια ε, πώς να το πω ακριβώς, ε, ε πώς εργάζεται το Κοινοβούλιο. Εμείς εξεργαζόμαστε στις νομοθετικές πράξεις, διαδικασία η νομοθετική και το Συμβούλιο κάνει τη δική του δουλειά. Ε, θα σας στηρίξουμε στην ειδική σας έκθεση ε, και πιστεύω ότι στην πλευρά του Συμβουλίου εκεί πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Ε, εμείς θα σας υποστηρίξουμε διότι έχουν οι πολίτες της Ένωσης το δικαίωμα να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν γιατί λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί προωθείται η συγκεκριμένη νομοθεσία σε κάθε περίπτωση και ενώ εμείς ε, ε, είμαστε γνωστοί, υπάρχουν τα τηλέφωνά μας, οι ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις, τα πρόσωπά μας, το Συμβούλιο είναι λίγο αδιαφανές, ένα black box. Η Άγχελα Βαλίνα. Ε, ευχαριστώ, καλημέρα, ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να πω, πέραν του να ευχαριστήσω και εγώ την Διαμεσολαβήτρια για το έργο που τελεί όλα αυτά τα χρόνια για να είναι μια πιο διαφανής Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή και σίγουρα για την αντιμετώπιση ενός πολύ σημαντικού προβλήματος που είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Από την ομάδα μας έχετε πλήρη υποστήριξη, την ΚΟΕ, e, αλλά θέλω και κάτι ακόμη να πω Σίγουρα υπήρξε σημαντική πρόοδος. Μην ξεχάσετε στην προσεχή έκθεση την επιτάχυνση και τη βελτίωση της ποιότητας των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στα έγγραφα αξιολόγηση που καταρτίζει, διότι συνηθίζει να αργεί πάρα πολύ με αυτά τα έγγραφα, όπως για παράδειγμα αναθεώρηση της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Και αυτό πρέπει να το διεκδικήσετε από την Κομισιόν, πιστεύω. Επίσης, έλλειψη πληροφοριών ε, σε ό,τι αφορά ε, τους εμπειρογνώμονες. Το λέμε από την αρχή της ε, θητείας και δεν αλλάζουν τα πράγματα. Επίσης, φυσικά η προστασία των πλέον ευάλωτων, των μεταναστών, και των προσφύγων, πρόθεση των διαδικασιών γρήγορης εκπαιρέωσης ε, και παροχής ασύλου. Αυτά είναι οι τομείς που μας ενδιαφέρουν και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Τζουτ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και από τη δική μου πλευρά. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει μια ευρεία συζήτηση για τη λογοδοσία του Συμβουλίου και την ειδική έκθεση. Αυτό είναι σημαντικό, πραγματικά. Και από την οπτική γωνία μιας βουλευτού που βλέπει την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, σίγουρα ε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαφάνεια και από τη συμπεριφορά του Συμβουλίου. Δεν είναι αρκετά εύκολο να δει κανείς πώς λαμβάνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η διαφάνεια, η λογοδοσία είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να θα επιτρέψουν μάλλον στους πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους. Ε, και σίγουρα ευθύνη μεγάλη έχει το Συμβούλιο και θα πρέπει να αναβαθμίσει ε, ε, τον τρόπο εργασίας του. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα παραδείγματα που μας δώσατε ε, για τις μη αμοιβόμενες περιόδους άσκησης. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και γνωρίζω ότι υπάρχει ένα intergroup στο Κοινοβούλιο που έχει προωθήσει μια εκστρατεία για την κατάργηση αυτών των μη αμοιβόμενων περιόδων άσκησης ε, στα γραφεία, παραδείγματος χάρη των Ευρωβουλευτών. Και ελπίζω να υπάρξει συνεργασία μεταξύ βουλευτών ε, και του δικού σας γραφείου γιατί πραγματικά πρέπει να πάψει εκμετάλλευση των νέων που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ε, εργαζόμενοι σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο όμως πέφτουν όλοι θύμα εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ Τζούντ, λέει πρόεδρος. Ακριβώς αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου, ότι δηλαδή αυτό που βλέπουμε και η Επιτροπή μας το συζητήσαμε μόλις πριν ναι, μεταξύ των συντονιστών. Έχουμε την σε ε, συμβάση πολύ δύσκολους όρου ε, ε, στη συμβάση εργασίας που πραγματικά επιφέρουν πλήγματα στην αξιοπρέπεια των ε, νέων και γενικώ των εργαζομένων. Επίσης ένας πολύ καλός ε, τομέας που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι ε, η αντιμετώπιση ακριβώς αυτής της επισφάλειας. Επίσης και για τη διαφάνεια πραγματικά κρατήστε ψηλά τη δάδα και θα συνεχίσετε το καλό έργο. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση που μας παρουσιάσατε. Πιστεύω ότι αυτό το βραβείο σας απονεμήθη ήταν πάρα πολύ, ε, ήταν κάτι που το αξίζατε πραγματικά πολύ και περιμένω με ουσία να σας ξαναδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, αν έχετε, ορίστε παρακαλώ. Κυρία Οράιλ, θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους Πραγματικά είναι ενθαρρυντικό πάντοτε να ακούει κανείς ενθαρρυντικά λόγια και λόγια υποστήριξης. Ε, κάποια από τα σχόλια Ιδίω αυτά που είπατε για το Συμβούλιο, την ειδική έκθεση για το Συμβούλιο, πραγματικά είναι ε, τόσο εύστοχα, γιατί ακριβώ αφορούν την ουσία αυτού που κάνουμε. Χωρίς σωστή ενημέρωση, ε, το αφήγημα, ε, το τελείως εσφαλμένο, δεν θα είχε οδηγήσει σε αυτές τις τόσο σημαντικές επιπτώσεις στην περίπτωση του δημοψηφίσματο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ελπίζω να έχω και στο μέλλον την υποστήριξή σας, όπως την έχω μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι. And now, colleagues, time has... συνάδελφοι, Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, αναφορά αριθμός 0143, εξ ονόματος ε, της πόλης του Μιλάνου για τη μετεγκατάσταση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στο Άμστερνταμ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να καλωσορίσω τον Δήμαρχο του Μιλάνου εδώ στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ, κύριε Δήμαρχε, με την ιδιότητα του αναφέροντα και για τη δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε μαζί σας. Πολύ εξημών έχουμε επισκεφθεί το Μιλάνο, μια πολύ όμορφη πόλη. Και θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσουμε την δική σας την άποψη όσον αφορά την μετεγκατάσταση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Προσβλέπουμε λοιπόν στην παρέμβασή σας έχετε το λόγο για μέγιστο 5 λεπτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να είμαι εδώ πέρα σήμερα, αξιότιμοι βουλευτές. Δεν είμαι εδώ πέρα σήμερα για να απαγγείλω κατηγορίες, αλλά από την άλλη δεν είναι τυπική και αόριστη παρουσία μου εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζει πραγματικά τι συνέβη και ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την υγεία των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Διαθέτει φάρμακα στην ευρωπαϊκή αγορά, η έγκαιρη διάθεση των οποίων μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις ζωές των πολιτών ή ακόμα και το καθεστώς επαγρύπνησης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ο βασικός στόχος της διαδικασίας της μετεγκατάστασης, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε από τον κανονισμό που εγκρίθηκε στις 22 Ιουνίου του 2017, είναι να συνεχιστεί η επιχειρηματική λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ο βασικός άξονας προκειμένου να έχουμε την επιχειρηματική αυτή συνέχεια προβλέπεται από τον ίδιο τον κανονισμό μέσω της άμεσης ε, διαθεσιμότητας ενός κτηρίου που θα έχει πολύ συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να διεκπερώνεται σωστά εργασία της EMA. Εμείς ε, ήδη από την αρχή είχαμε λάβει κάποιες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν θα έπρεπε να κατασκευάσουμε νέα ad hoc κτίρια που θα οδηγούσαν ουσιαστικά σε δύο διαδοχικές μετακομίσεις γιατί δεν θα προβλεπόταν ο απαραίτητος χρόνος για κάτι τέτοιο ούτε θα έπρεπε να κτιστεί εκ νέου ένα κτίριο, γιατί αυτό ενδεχομένως να έθετε εν κινδύνο την ίδια την συνέχεια της λειτουργίας της υπηρεσίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ακριβώς επειδή στο Μιλάνο είχαμε τον απαραίτητο χρόνο, χώρο με συγχωρείτε, εξ αρχής τηρήσαμε τις ενδείξεις αυτές και χάρη στην πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με την περιφέρεια της Λομβαρδίας, επιλέξαμε ένα κτίριο μεγάλης ερτεκτονικής αξίας, ιδιαίτερα λειτουργικό, που βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης. Ο ουρανοξύστης Πιρέλη όντως παρέχει τους κατάλληλους χώρους, μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν, βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, σε ένα από τα σημεία με πάρα πολύ καλές άλλες διασυνδέσεις. Περιμέναμε λοιπόν ότι τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά της Ιταλικής υποψηφιότητας θα λαμβάνονταν πολύ σοβαρά υπόψη στα πλαίσια της απόφασης για τη νέα έδρα της υπηρεσίας, σύμφωνα πάντα με μια διαδικασία, με μια διαδικασία διαφανούς αξιολόγησης και λήψης απόφασης, μιας διαδικασίας που θα ήταν πραγματικά αξιοκρατική. Δεδομένου επίσης, δεδομένης επίσης όλες αυτές τις που χρειάστηκε να κάνουμε για να καταρτήσουμε αυτόν τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητα. Όπως ξέρετε, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 20 Νοεμβρίου 2017 ελήφθη απόφαση βάσει της οποίας το Μιλάνο έλαβε τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη και στη δεύτερη ψηφοφορία. Μετά την τρίτη ψηφοφορία δημιουργήθηκε μια κατάσταση ισοψηφίας και είδαμε αμέσως ότι προχωρήσαμε σε μία κλήρωση και κλεισμένων των θυρών χωρίς καμία απόλυτος διαφάνεια με την άμεση καταστροφή όλων των ψηφοδελτίων που είχαν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες πληροφορίες και χωρίς να συνταχθούν καθόλου πρακτικά. Επίσης βλέπουμε ότι ενώ κατά τη διάρκεια των πρωινών εργασιών ήταν ανοιχτή η λεγόμενη αίθουσα ακρόαση, κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία αλλά και τη κλήρωση η αίθουσα αυτή έκλεισε και κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επαλήθευση τη όλη διαδικασία και προφανώ καμία απολύτω διαφάνεια. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα άλλο προ αυτό. Πάντω η αρχική μα έκπληξη για την ακολουθητή αυτή διαδικασία αυξήθηκε ακόμα περισσότερο όταν μάθαμε ότι η πόλη η οποία επελέγει τελικά για κλεισμένο των θυρών και μέσω κλήρωσης δεν είχε τελικά το κατάλληλο κτίριο να προτείνει και πρότεινε την μετακόμιση σε μια προσωρινή και έπειτα την κατασκευή ενός καινούριου κτίριου. Επίσης η κυβέρνηση της πόλης αυτής ακολουθώντας μια παράτυπη διαδικασία, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκρύψει το τμήμα εκείνο της υποψηφιότητάς της που είχε να κάνει με την μεταβατική έδρα, την προσωρινή έδρα. Υπάρχουν όμως δύο ακόμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Τον Ιανουάριο του 2018 φάνηκε ότι και η μεταβατική έδρα που πρότεινε η επιλεγήσα και οι δύο μεταβατικές έδρες που πρότεινε η επιλεγήσα τελικά πόλη ήταν ακατάλληλες και αυτό το έκρινε η ίδια η αίμα και ότι θα πετούσαν τελικά πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερα έξοδα για να προσαρμοστούν οι δύο αυτές έδρες και για να κτιστεί το νέο κτίριο. Επίσης βλέπουμε ότι μετά την ψηφοφορία τροποποιήθηκαν διάφορα στοιχεία του αρχικού φακέλου του Άμστερνταμ και καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά βάλει κατά τη ίση μεταχείριση και τη διαφάνεια. Για όλου αυτού του λόγου, εμεί αποφασίσαμε να κάνουμε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε τώρα καθυστέρηση σε σχέση με την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία και γνωρίζουμε ότι θα έπρεπε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 2019 τελικά να είναι έτοιμο το νέο αυτοκτήριο κτίριο προτείνει το Άμστερνταμ. Αν καθυστερήσουμε τόσο πολύ θα, θα ζημιώσουμε τους ίδιους Ευρωπαίους πολίτες. Και πρέπει να γνωρίσουμε επίσης και ποιες είναι οι πραγματικές δαπάνες της προσωρινής μετακόμισης και της μόνιμης έπειτα μετακόμισης στο Άμστερνταμ. Εμείς στην υποψηφιότητα του Μιλάνου δώσαμε όλα τα ακριβή στοιχεία και για το ενίκιο και για τα γενικότερα ποσά και τις υπόλοιπες δαπάνες που θα έπρεπε τέλο πάντων να ληφθούν για να γίνει μετακόμιση αυτή 59 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα. Αντίθετα, στο παράρτημα τη υποψηφιότητα στο Άμστερνταμ γίνεται μία αναφορά σε μία φορολογική διευκόλυνση 18 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς όμως να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά την πραγματική μίσθωση του κτηρίου που θα αποτελέσει τη νέα έδρα της, του Άμστερνταμ, τη υπηρεσία αυτής τη EMA. Επομένω, εμεί ζητάμε τρία πράγματα αυτή τη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτον, να διασφαλίσετε μια πάρα πολύ αυστηρή παρακολούθηση, μια αποτελεσματική παρακολούθηση της όλης διαδικασίας μετακόμισης, ιδίως όσον αφορά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η πρότασή μας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβλέψει μια κάποια εφεδρική, εναλλακτική αν θέλετε λύση και για μας η εναλλακτική λύση δεν είναι άλλη παρά η πρόταση του Μιλάνου. Δεύτερον, σας ζητούμε να αποτιμήσετε το πραγματικό κόστος μετακόμισης της υπηρεσίας στο Άμστερνταμ και τρίτον, να κρατήσετε ανοιχτή τη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου και να λάβετε υπόψη επίσης και την όλη δικαστική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Το Μιλάνο αξιότιμοι ευρωβουλευτές όχι μόνο παρουσίασε μία πλήρη υποψηφιότητα, αλλά επίσης έδειξε ότι ήταν σε θέση το κατάλληλο χρονικό διάστημα να υποδεχθεί την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ε, έχουμε μαζί μας ε, σήμερα την μόνιμη, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Τζοβάνι Πουλιέζερ το μόνιμο αντιπρόσωπο στα ευρωπαϊκά όργανα. Έχετε το λόγο για το πολύ δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Δεν χρειάζομαι καν δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ εμείς έχουμε υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Μιλάνου ως Ιταλική κυβέρνηση για την αίμα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η πόλη αυτή τη Λομβαρδίας είναι σε θέση να διασφαλίσει την απόλυτη και αποτελεσματική συνέχιση των εργασιών της αίμα που θα φύγει 31 Μαρτίου 2019 από την Βρετανία. Για την Ιταλική υποψηφιότητα υπενθυμίζω ότι υπάρχει ήδη χώρος λειτουργικός, ε, κρατικός, απόλυτα προσαρμόσιμος σε χρόνο γρήγορο για τις απαιτήσει της ΕΜΑ και του προσωπικού του. Η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης αφού προέκυψαν στοιχεία ε, για ε, λήψεις ε, της Ολλανδικής προσφοράς και χρονικά και ε, απόψη κόστους. Εμείς λοιπόν είχαμε στόχο να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της λειτουργίας της ΕΜΑ για τη διασφάλιση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονό ότι οι δράσεις της Ιταλικής κυβέρνησης έφεραν ε, τη διόρθωση ορισμένων ε, πτυχών που δεν συμμορφώνονταν ε, με την προσφορά. Σε αυτά αναφέρθηκε το Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο για την προσφορά του Άμστερνταμ. Παρότι απομένουν αμφιβολίες κατά πόσο μπορεί η Ολλανδία να τηρήσει αυτά που υποσχέθηκε ειδικότερα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της νέας έδρας. Συμπερασματικά, κυρία Πρόεδρε, εμεί ε, ω Ιταλική Κυβέρνηση υποστηρίζουμε απόλυτα το Δήμο του Μιλάνου και τη δυνατότητά του να φιλοξενήσει την ΕΜΑ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Χίλια ευχαριστώ στα Ιταλικά. Έχει έρθει η ώρα να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν, τον κύριο Κλάου. Δεν βλέπω που βρίσκεται. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. I would first of all like to state that the και ευχαριστώ τους αναφερόμενους. Θέλω να πω ότι η Κομισιόν θεωρώ ότι τέτοιες καταγγελίες ε, δεν στρέφονται κατά της Κομισιόν αλλά κατά των διαδικασιών του Συμβουλίου. Εκεί πρέπει να στραφούν. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό σε ένα λεπτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ε, ποια είναι το πλαίσιο της συζήτησης αυτής. Με πλαίσιο ότι εννοώ ότι σήμερα. Έχουμε συγγενείς του προσωπικού της ΕΜΑ που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή να μετεγκατασταθεί από το Λονδινό στο Άμστερνταμ ε, το καλοκαίρι ήδη ώστε να είναι έτοιμοι για το επόμενο σχολικό έτος. Επίσης βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης της νομοθετικής πρότασης ε, για τον κανονισμό αίμα που θα επιβεβαιώνει τη μελλοντική έδρα και την ημερομηνία με Επίσης, Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία για το κτίριο, όπως την ονομάζουμε, μιλάμε για το Άμστερνταμ, όπου οι δημοσιονομικές αρχές, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχουν ήδη εγκρίνει το έγγραφο για το κτίριο που υπέβαλαν οι Ολλανδικές αρχές. Το ότι τα λέμε όλα αυτά δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν ε, υιοθετεί κάποια θέση υπέρ των κατοχωρών και του Άμστερνταμ και κατά οποιασδήποτε άλλη αίτηση, η Κομισιόν και θέλω να το υπενθυμίσω αυτό παρότι κανονικά θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι δεν διαδραμάτισε κανέναν επίσημο ρόλο στη λήψη αυτή τη απόφαση. Τι έκανε όμω η Κομισιόν ότι βάσει τη διαδικασία, η οποία στις 22 όπω είπε πολύ σωστά ο, Δήμαρχο ο δήμαρχος του Ιουνίου πέρυσι εγκρίθηκε η διαδικασία σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, όχι από αξιωματούχου. Και βάσει αυτή της διαδικασίας η Κομισιόν διεξήγαγε μια αξιολόγηση βάσει κριτηρίων που είχαν διατυπωθεί στη διαδικασία αυτήν. Η αξιολόγηση αυτή δεν κατέληξε σε οποιαδήποτε σύσταση, σε καμία λίστα επιλαχόντων, σε καμία κατάταξη. Η Κομισιόν απλά έδωσε στοιχεία, πληροφορίες βάσει των προσφορών που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη, αυτά που συμμετείχαν στη διαδικασία. Και με πολύ απλό, νυφάλιο τρόπο παρήχε η Επιτροπή αυτές τις πληροφορίες στα 27 κράτη-μέλη, τα οποία τον Νοέμβριο πέρυσι το φθινόπωρο έλαβαν την τελική απόφαση. Όπως λέω λοιπόν δεν υπερασπίζομαι την επιλογή την τελική απόφαση. Απλά να σας υπενθυμίσω αυτό που υπόθηκε και στη διαδικασία. Λέγεται ότι η απόφαση θα λαμβάνεται με μια διαδικασία ψηφοφορίας που βρίσκεται στο κεφαλαίο 6 πιο κάτω στη διαδικασία η έκβαση της οποίας θα βρίσκει σύμφωνα τα κράτη-μέλη όπως συμφωνούν τα κράτη-μέλη εκ των προτέρων. Δηλαδή η διαδικασία είχε συμφωνηθεί, είχε συζητηθεί, είχε προετοιμαστεί επαρκώς από τα κράτη-μέλη και από τα 27 μήνες πριν. Όταν τα κράτη-μέλη υπέβαλαν Ετήσεις τέλη Ιουλίου υπήρχε πάρα πολύς χρόνος, άφθονος χρόνος για συζήτηση. Τα κράτη-μέλη που υπέβαλαν προσφορέ ε, είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσει. Τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο, να ζητήσουν εξηγήσει. Υπήρχε άφθονο χρόνο για εξηγήσει ε, και για διευκρινήσει πριν λάβει η χώρα η ψηφοφορία αυτή καθεαυτή τον Νοέμβριο. Εγώ δεν θέλω να εκφέρω οποιαδήποτε άποψη όσον αφορά τη διεξαγωγή τη ψηφοφορία γιατί αποτελεί απόλυτη αρμοδιότητα του, του Συμβουλίου. Συγγνώμη. Αλλά ένα πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, φυσικά ήταν μία διαδικασία που γίνεται μία φορά που, αφορούσε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είχαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε ε, ξανά τέτοια περίπτωση όπου ένας-δυο οργανισμοί ε, πρέπει να αποφασιστεί πού θα βρίσκονται που θα μεταφερθούν και όπου είχαμε 27 προσφορές γι' αυτό. Οπότε αυτή η διαδικασία ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και ούτε αποτελεί προηγούμενο για μελλοντικέ διαδικασίες καθορισμού έδρας οργανισμών. Οπότε στη διαδικασία αυτή έπρεπε να διασφαλίζεται ότι στο πέρας της διαδικασίας θα, θα, θα, θα καταλήγαμε όλοι σε κάποια απόφαση θα υπήρχε κάποια απόφαση και μαθηματικά όπως καταλαβαίνετε και στις δύο περιπτώσεις ε, αυτό ε, που έγινε δεν το περίμενε κανένας. Οι δύο συναγωνιστές ε, έλαβαν υποψηφία μετά από το δεύτερο γύρο. Κανείς δεν το περίμενε αυτό και στην ΕΜΑ και στην ΕΜΑ. Ναι, και το να τραβήξουμε κλήρο δεν ήταν κάτι που ήθελε κανένας Ναι, συμφωνώ, αλλά υπήρχε ήδη στη διαδικασία από τον Ιούνιο, οπότε δεν έπρεπε να εκπλήξει κανέναν. Ήταν κάτι που είχε θεσπιστεί και το είχαν δεχτεί όλοι ότι αυτή θα ήταν η διαδικασία σε περίπτωση ισοψηφία. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας διαβεβαιώ όμως ότι ο αναφέρον και η ομάδα του Μάλλον λέω προ τον αναφέροντα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρώτη φορά ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει τόσο παθιασμένα. Σίγουρα προηγούμενο τέτοιο δεν είχαμε στο παρελθόν. Η κατάσταση όντω είναι πολύ περίεργη ασυνήθιστη και νομίζω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι δεν ξέρανε τελικά πάρα πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν, πώς έπρεπε να κινηθούν στο μέλλον κτλ. Πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε τώρα, ας ακούσουμε τους συναδέλφους. Η Ελενόρα Εύη πρώτη. Μέγιστο δύο λεπτά, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. έχοντας ακούσει την παρέμβαση του Δημάρχου του Μιλάνου, του κυρίου Σάλα, τον οποίο πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ που παρουσίασε την αναφορά αυτή και που έχοντας ακούσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν συνεχεία, πραγματικά θα μπορούσα να πω ότι η αρχή της διαφάνειας, της δημοσίευσης, της διαδικασίας επιλογής όσον αφορά την διαδικασία κατάσταση των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά τέθησαν εν αμφιβόλο. Νομίζω ότι πραγματικά το τέχνασμα αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε, να ληφθεί δηλαδή μια τόσο σημαντική απόφαση στο περιθώριο ενός Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικά είναι κάτι το οποίο καταγγέλουμε, είναι αξιολύπητο πραγματικά. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έρχεται στις συνοδευτικές εκθέσεις για την πρόταση κανονισμού που τροποποιεί τον προηγούμενο κανονισμό όσον αφορά την EMA, η ίδια έρχεται και λέει ότι ε, η μετεγκατάσταση της έδρας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Από την άλλη βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φρόντισε καθόλου να εμπλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετέθη εντελώς στο περιθώριο της όλης διαδικασίας και προφανώς εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το δεχτούμε στο μέλλον. Επίση σε μια τόσο σημαντική απόφαση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζημιώνεται και η ίδια η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός αυτός των φαρμάκων, όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και όσον αφορά και το δημοσιονομικό σκέλος, γιατί η απόφαση που ελήφθη θα βαρύνει και τις τσέπες, όχι μόνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Επομένω, έχω την εντύπωση ότι ακόμα και στην πρόταση την τροποποιητική για τον κανονισμό όσον αφορά τον νέο Αυτοευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον. Θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η πρακτική πάση θυσία. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως η δική μας Επιτροπή Αναφορών να αποστείλει μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο, αλλά κυρίω στους επικεφαλείς διαπραγματεύσεων για τον τριμερή διάλογο του EMA και να τους ζητήσουμε να λάβουν υπόψη τους προφανώς τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο, ας μην το ξεχνάμε, ζήτησε να εμπλακεί στο μέλλον πλήρως στην όλη διαδικασία και ζήτησε επίσης να υπάρχει και μια εφεδρική λύση σε περίπτωση που το Άμστερνταμ τελικά δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του από άποψη κόστου και από άποψη χρόνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης η αναφορά αυτή να, ληφθεί, να παραμείνει ανοιχτή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλου του ευρωβουλευτέ να ενημερωθούν για το τι έγινε, να συλλέξουν σε απαραίτητε πληροφορίε και να περιμένουν επίση να δουν και ποια θα είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εκκρεμεί δικαστική απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου. Α μην το ξεχνάμε αυτό. Ο κύριος... Ευχαριστούμε, κύριο Τσίριο. Συγγνώμη, πάντα κάνω λάθο με αυτό το όνομα. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Δήμαρχο τον κύριο Σάλα και ευχαριστώ την Πρόεδρο που δέχθηκε το αίτημά μας να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό ω κατεπήγον. Εδώ δεν μιλάμε για την Ιταλία κατά των υπολείπων χωρών τη Ευρώπη, ούτε Μιλάνο κατά Άμστερνταμ ή άλλων πρωτευουσών. Εδώ μιλάμε για μια διαφορετική διαδικασία. Εμεί είμαστε στην Επιτροπή Αναφορών και πρέπει να καταλάβουμε αν η διαδικασία ε, καθορισμού της νέας έδρας της ΕΜΑ ε, τήρησε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί διαφάνειας, ε, και δικαιοσύνη. Γιατί αύριο μπορεί να είναι η Ρουμανία, η Ισπανία, κάποια άλλη χώρα. Αυτό είναι το καθήκον μα σήμερα και αυτό αποτελεί αντικείμενο σαφώ αυτή τη αναφορά. Αυτή η αναφορά δεν είναι να μπούμε επί τη ουσία να δούμε αν έπρεπε να διαλέξουμε τη μία έδρα ή την άλλη. Το θέμα είναι να δούμε, ε, ρωτώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρξε η διαφάνεια που θέλαμε, γιατί κοιτώντας τις διάφορες ενδείξεις που έχουμε ότι δεν υπήρξε διαφάνεια, είναι πολλές αυτές οι ενδείξεις. Το θεμα ειναι να δουμε ρωτώντα την ευρωπαικη επιτροπη υπηρξε η διαφανεια που θελαμε γιατι κοιτώντα τι διάφορε ενδείξει που εχουμε οτι δεν υπηρξε διαφανεια ειναι πολλέ αυτέ οι ενδείξει. το γεγονό οτι κατω χώρε αποφάσισαν το που θα έχει έδρα και που αυτό ήταν το αδύναμο σημείο της προσφοράς τους ε, ε, ουσιαστικά δεν το ανακοίνωσε το που θα βρισκόταν η έδρα και αυτό το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονός ότι έγιναν οι ψηφοφορίες χωρίς να υπάρχουν πρακτικά, το ότι η ακρόαση ε, έγινε με κλειστή την κάμερα όταν Χρειάστηκε. Εμεί θέλουμε, ξέρετε, οι Ευρωπαίοι πολίτε να πιστεύουν στην Ευρώπη. Από εγώ να πω στου Ευρωπαίου πολίτε ότι η Ευρώπη επέλεξε τη νέα έδρα τη ΕΜΑ ψηφίζοντα και μετά ε, τα ψηφοδέλτια, χωρί πρακτικά, ε, σβήνοντα την κάμερα. Ε, ξέρετε, εκεί χάνεται η αξιοπιστία τη Ευρώπη, ανεξάρτητα τη ΕΜΑ, ε, του Μιλάνου και του Άμστερνταμ. Γι' αυτό τον λόγο σήμερα στην Επιτροπή μα απαιτείται να υιοθετήσει μια θέση η Επιτροπή μας να κρατήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά να υπάρξει προσφυγή στο δικαστήριο γιατί μπορεί να γίνει με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και να παρακολουθήσουμε τι έγινε στην Ολλανδία. Δεν τίθε το ζήτημα εδώ Μιλάνο ή Άμστερνταμ, τίθε ε, ο ζήτημα η αμστερνταμ τιθε ο ζητημα η εξουπιστία της Ευρώπης μας. Ε, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπόλτζαν, καλώς ορίσατε. Ήσασταν κι εσείς μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, αν κατάλαβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί είμαι σύνδεσμος ε, από τον Οργανισμό Φαρμάκων ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι και σκιώδης εισηγήτρια της έκθεσης ε, για την κατάσταση του Οργανισμού Φαρμάκων. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που είπαν σήμερα ότι η διαδικασία αυτή του να γίνει κορώνα γράμματα δηλαδή για την απόφαση είναι προβληματικό. Υπάρχει δήλωση Συμβουλίου Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2012 που λέει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει για τι έδρε των ε, τελεστικών οργανισμών. Είναι προβληματικό λοιπόν αυτό που έγινε για εμάς. Ε, τώρα θέλω να τονίσω ότι η διαδικασία αποφασίστηκε από το Συμβούλιο δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, μήνες πριν την ψηφοφορία, και κανείς δεν είχε να πει τίποτα αντίθετα. Επειδή υπήρχαν ανησυχίε ό,τι αφορά την προσωρινή έδρα ε, στο Άμστερνταμ που δεν είναι επαρκή ε, και το σχέδιο του νέου κτηρίου μάλλον δεν θα έχει ολοκληρωθεί η ανήγερσή του έγκαιρο, ε, οργανώσαμε μια επίσκεψη. Επισκεφθήκαμε το Φεβρουάριο το Άμστερνταμ και ο διευθυντή του ΕΜΑ και εκπρόσωπο τη Ολλανδική κυβέρνηση ήταν εκεί και μα έδωσαν διαβεβαιώσεις. Είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια, υπάρχουν περιορισμοί και υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία του οργανισμού αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που ε, εγκρίθηκε το Άμστερνταμ, το να είναι δηλαδή ε, πιο ε, εύρυθμη λειτουργία. Καταλαβαίνω λοιπόν πώς νιώθουν οι πρόσωποι του Μιλάν και εγώ το ίδιο θα ένιωθα στη θέση σας. Εμείς επιβλέπουμε τα φάρμακα και δεν θα πρέπει η εργασία της να τεθεί σε κίνδυνο ε, εταιρεία του οργανισμού. Η πρώτη ψηφοφορία για τον οργανισμό περί ε, είχε ένα αποτέλεσμα μεγάλη πλειοψηφία. Προσωρινά δηλαδή επικυρώθηκε ως έδρα του οργανισμού του Άμστερνταμ με συγκεκριμένε προϋποθέσεων συγκεκριμένου όρου. Τώρα έχουν ξεκινήσει τριμερείς διάλογοι και ξεκαθαρίσαμε στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν ότι με την κατάσταση του αίμα ε, είναι η τελευταία φορά ε, που αναμένεται να βάλει απλά τη σφραγίδα του Κοινοβούλιο στο τέλος ε, εφόσον είναι συνομοθέτε, Δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια και εκτό τη διαδικασία. και πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση της κοινή δήλωση. Πώς λύνεται τώρα το πρόβλημα. Αυτό θα εξαρτηθεί από την έκπληξη των διαπραγματεύσεων σε μεγάλο βαθμό και ολοκληρώνοντα θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντλήσει τα διδάγματα των προβλημάτων που ανέκυψαν με την μετακατάσταση του οργανισμού φαρμάκων. Σίγουρα υπάρχουν λάθη που στο μέλλον θα πρέπει να αποφευχθούν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και για τη συμβολή σα που πραγματικά ήταν πάρα πολύ πολύτιμη αυτή τη χρονική στιγμή. Είναι σημαντικό και για του αναφέροντε να το γνωρίζουν δηλαδή ότι γίνονται αυτή τη στιγμή οι τεμερεί διάλογοι. Ο ένα έχει ολοκληρωθεί και προβλέπεται και έτερο ε, άμεσα. Επίση ε, είναι και καλό εισηγητή από την Επιτροπή Αναφορών, κύριο ε, Λαβία. Να πάμε στην κυρία Άουκεν, την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Εγώ είμαι από την Κοπενχάγη, που ήταν υπαριθμόν τρία πόλη σε διαδικασία, όπως υποψήφετε. Και εμείς νιώσαμε προσβεβλημένοι και είμαι σίγουρη ότι και η η κυβέρνηση ε, ήταν εξίσου εξαρτησμένη με την Ιταλική που δεν συμμετείχε το κοινοβούλιο ή που δεν υπήρχε διαφάνεια. Διαμαρτυρήθηκε όμως καμιά κυβέρνηση. Όχι ούτε η Δανέζικη ούτε η Ιταλική. Τα βρήκαν όλα τέλεια που το κοινοβούλιο ήταν απ' έξω. Το βρήκαν δίκαιο που δεν υπήρχε διαφάνεια. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η αρρώστια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η παθογένεια, το Συμβούλιο να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν να είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός και όχι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και νομίζω ότι η διαδικασία με τη μετακατάσταση της έδρας στο αίμα ε, ε ήταν μια ε, πολύ εύγλωτη περίπτωση του πόσο προβληματική είναι η κατάσταση. Αλλά πραγματικά είναι λυπηρό ε, να ε, διαμαρτύρονται και να διαρρύνουν τα αίματιά τους αυτοί που δεν διαμαρτυρήθηκαν καθόλου στην αρχή. Γιατί υπάρχει αυτό το απόρριτο και τα διακυβερνητικά χουνέρια και συνεχίζονται αυτά. Στην Επιτροπή ΕΝΒΗ υπάρχει αυτή η διαδικασία τώρα που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν που το λέω, αλλά θα λήξει σύντομα αυτή η διαδικασία. Ήμουν σαν προσωπικό που πήγε στο Άμστερνταμ. Αυτά που είδαμε και ακούσαμε εκεί ήταν πιστικά, οφείλω να πω. Δεν λέω ότι δεν θα ήταν το ίδιο με το Μιλάνο. Αλλά αυτά τα είδαμε στο Άμστερνταμ. Και ήταν και αυστηρές προποθέσεις που μπήκαν στην νομοθεσία για το χρονοδιάγραμμα, οικονομικές προποθέσεις. Υποτίθεται ότι θα τηρηθούν όλα από το Άμστερνταμ και δεν θα υπάρχει κανένα κενό και παραθυράκι. Σα το υπόσχομαι. Σίγουρα βοηθάει πολύ που είστε εδώ για να καταλάβουν όλοι ότι η προσοχή μα είναι πλήρω στραμμένη στο τι συμβαίνει εκεί. Και ελπίζω και στο μέλλον η Ιταλία να είναι στο πλευρό μα, στο πλευρό του Κοινοβουλίου. Ώστε το Συμβούλιο είναι πολύ πιο ανοιχτό να συμμετέχει και να ε, δίνει συμμετοχή όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Κοινοβούλιο πάντως το Ευρωπαϊκό σίγουρα πρέπει να συμμετέχει σε τις διαδικασίες αυτές. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά και ελπίζω να αλλάξει η νοοτροπία και με τη δική σας βοήθεια. Ευχαριστούμε κύριε Σκοσολίνο. Η πρώτη συζήτηση είχε ολοκληρωθεί τώρα. Ας παραμείνουμε στα γεγονότα να σταθούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε επίσης. Εγώ θα ζητούσα από την Πρόεδρο να διατηρήσει ανοιχτή την αναφορά και αυτό είναι το ελάχιστο αυτή τη στιγμή. Να μην κάνει λοιπόν μόνο αυτό, αλλά να μας ενημερώνει μέσα στους επόμενους δύο-τρεις μήνες, όχι παραπάνω, ώστε να μαθαίνουμε τι γίνεται με την κατάσταση. Ας ανακτήσουμε, αν μπορούμε, μια πλήρη, ε, τον πλήρη ρόλο του Κοινοβουλίου, βήμα προς βήμα, για να δούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Κατά την άποψή μου, η Κομισιόν μας είπε διάφορα πράγματα. Τι να σας πω. Εσείς ξέρετε ότι η Ιταλική κυβέρνηση έθεσε βέτο στην πρώτη φάση της διαδικασίας, το οποίο ήρε στη συνέχεια το Συμβούλιο όταν ανέλαβε πλήρη ευθύνη η Κομισιόν για τις αποφάσεις. Και η δική μου στάση, εντάξει μπορεί να είναι δική μου προσωπική στάση, δεν θέλω να πω ότι είναι και άλλον. ήταν ότι η Κομισιόν έπρεπε να ενημερώσει το Συμβούλιο ότι δεν ήταν ίσες οι τρεις προτάσεις. Άλλο είναι να προτείνεις ένα κτίριο το οποίο λειτουργεί πλήρως ήδη, άλλο είναι να προτείνεις ένα κτίριο το οποίο πρόκειται να οικοδομηθεί. Δεν είναι ίδια η απόφαση λοιπόν. Δεν είναι ισότιμες επιλογές, είναι δύο επιλογές εντελώς διαφορετικές και το Μιλάνο θα μπορούσε να προσφέρει κάτι άλλο. Για τη διαδικασία λοιπόν εντάξει θα μπορούμε να συζητάμε πάπυρον για το παραδεκτό της ε, ε, διαδικασίας αυτής. Το θέμα είναι ότι καταλήξαμε κάπου δύο όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αναμφίβολα το Άμστερνταμ υπέβαλε μία πρόταση εντελώς διαφορετική από αυτή του Μιλάνου. Άλλο είναι να προσφέρεις ένα κτίριο ήδη που υπάρχει ήδη και άλλο είναι να προσφέρεις ε, τη δυνατότητα να οικοδομηθεί ένα κτίριο. Οπότε ας παραμείνουμε στα γεγονότα, ας παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις διότι αφορά τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και ας ε, παραμείνουμε ενήμεροι με στους επόμενους μήνες, ας μείνουμε σε επαφή ώστε να δούμε τι γίνεται με την οικοδόμηση του χώρου στο Άμστερνταμ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά τελειώνει ο χρόνος. Σε λίγο δεν θα έχουμε διερμηνία. Πέτερ Γιάρα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και του αναφέροντες πολύ σύντομα. Τρία είναι τα προβλήματα που βλέπω εγώ. Το πρώτο συμμετοχή του κοινοβουλίου ναι ή όχι στο μέλλον. Αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για το μέλλον βέβαια. Όταν θα ξανασυζητήσουμε τέτοια θέματα. Το δεύτερο που με ανησυχεί. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού όσο παίζεται το παιχνίδι. Μπορούμε να έχουμε κάποιες απαιτήσει ε, και δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να καταλήξουμε ε, σε ε, διάφορες συγκρίσεις και να πούμε αυτό μπορούσε να γίνει, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Και το τρίτο, το Άμστερνταμ το έχει πλέον φαίνεται εξασφαλίσει το θέμα. Τώρα το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι όμως ποιος ελέγχει ε, όταν υπάρχουν κάποια κριτήρια παραδοσιακά τα οποία ορίζονται από την Κομισιόν. Ποιο εγγυάται ότι τηρούνται και λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, ε, αν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και απαιτήσει ε, που τελικά μετά δεν τηρούνται, στην Πρέψη για παράδειγμα, ποιος φέρει την ευθύνη, τι γίνεται εκεί. Αυτά πρέπει να τα λέμε πίσω υπόψη και είναι σημαντικό να υπάρχει fair play. Ευχαριστούμε πολύ. Μας δείξατε κι εσείς ότι μπορεί να είναι κανείς συγκεκριμένο και σύντομος. Ο κύριος Πεντιτσίνη τώρα έχει το λόγο. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ είμαι μέλος της ε, Επιτροπής ε, που ασχολείται με τις διαπραγματεύσει ε, για την αίμα. Συμμετέχω επίσης και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν πριν από λίγο. Όντως, η Ολλανδική υποψηφιότητα, η Ολλανδική προσφορά ήταν τελικά διαφορετική στην πράξη από αυτή που παρουσίασαν αρχικά οι Ολλανδικές αρχές. Η προσφορά που αξιολόγησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε να κάνει με μια άλλη προσφορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί η ρήτρα εμπιστευτικότητα που ζήτησαν και απέτησαν οι Ολλανδικές αρχές ουσιαστικά έγινε αποδεικτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εν συνεχεία ανακάλυψε την πραγματική προσφορά της Ολλανδίας, είπε ο ίδιος οργανισμός ότι δεν ήταν επαρκής αυτή η προσφορά, δεν ήταν κατάλληλη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Τώρα, χρησιμοποιήθηκε κλήρωση, καταλήξαμε στη νέα αυτή προσφορά που εγκρίθηκε τελικά και η οποία τελικά τι περιέχει. Μία μεταβατική ουσιαστικά λύση, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η μίσθωση μιας προσωρινής έδρας μέχρι να οικοδομηθεί ένα νέο κτίριο και ότι εκεί πέρα ουσιαστικά θα μπουν οι κύριες λειτουργίες, οι βασικές μονάδες της ΣΕΜΑ, ενώ στο μόνιμο κτίριο το οποίο θα οικοδομηθεί στο μέλλον θα τοποθετηθούν, θα τοποθετηθούν οι υπόλοιπε. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό θέτει εν κινδύνο την όλη λειτουργία του οργανισμού. Αν υπάρξει οποιαδήποτε νομικό ή τεχνικό πρόβλημα, αυτό σε θα θέσει εν κινδύνο τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει όντως η δική μας η Επιτροπή να αποστείλει μία επιστολή που θα ζητά να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και θα πρέπει επίσης να έχουμε και τη συνεισφορά της Ιταλικής κυβέρνησης αλλά και, της, ε, του Δήμου του Μιλάνου. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πατρίτσια Τόια έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι μιλώ ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το λέω στη φίλη και στην Αλφα δεν είμαστε εδώ Ιταλοί βουλευτέ. Είμαστε ευρωβουλευτέ. Ε, Μα ενδιαφέρει να υπερασπίσουμε τα προνόμια του Κοινοβουλίου, τα οποία συνέθλεψαν αυτή τη στιγμή. Δεν τα έλαβε κανεί υπόψη. Είναι απαγορεύεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Πρέπει να το καταγγέλουμε. Ω ευρωβουλευτέ είχα να πω αυτό. Το δεύτερο με ανισχύει ο ρόλο τη ε, Κομισιόν. Πολύ ειλικρινά το λέω στον εκπρόσωπο Τη ε, Κομισιόν. Κάθε φορά με άλλο συνομιλητή έχουμε. Δεν υπήρξε διαφάνεια ούτε σαφήνεια στα έγγραφα. Δεν μα τα έδωσε κανεί όταν τα ζητήσαμε εκ των υστέρων μετά από την επιλογή. Δεν μα έδωσε κανεί. Απαντήσει, ε, Λάβαμε προσβολέ ε, όσον αφορά την ιδιότητά μα και δεν καταλαβαίνουμε ποιο έγγραφο, ποιο ρόλο παίξατε, ποιο ρόλο έπαιξε ποιο. Σα κάνω μια ερώτηση. Όσον αφορά την αξιολόγηση τη Ολλανδική πρόταση, σε ποια έγγραφα βασιστήκατε, βάσει ποια πρόταση, τη πρώτη, τη δεύτερη, ποια δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Σε αυτή την Ευρώπη που υποτίθεται ότι είναι διαφανή, εμά δεν μα αρέσει, σε εμά του φιλευρωπαϊστέ, τέτοια έλλειψη διαφάνεια. Το τελευταίο, ω μέλο του Κοινοβουλίου και ω Ευρωπαία πολίτη, ανησυχώ ότι αυτό το σοφάκελο αντίκειται στα συμφέροντα των πολιτών για τη φαρμακοπαγρύπνηση, για τα νόβα φάρμακα. Αν ξεσπάσει κάποια επιδημία και εμεί δεν είμαστε έτοιμοι, ποιο θα φέρει την ευθύνη. Πρέπει να διασφαλίσουμε και στα, σας και εκλυπαρώ κυρία Πρόεδρε. Ας διατηρήσουμε ανοιχτό το φάκελο. Ας βάλουμε μια προθεσμία, δύο-τρεις μήνες, να παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε σημαίνει θέλω να ξέρω ποιος παρακολουθεί, τι στοιχεία συγκεντρώνει, ποιος ελέγχει, τι, ποιον ελέγχει, αυτός που ελέγχει, πώς συνεχίζεται η διαδικασία. Και τέλος να έχουμε και ένα εφεδρικό σχέδιο. Ε, πάντα κάνουμε κρυφά σχέδια ας έχουμε και ένα εφεδρικό Μιλάνο, κοπενχάγη κάτι, ένα recovery plan, συγγνώμη, όχι μυστικό σχέδιο, ένα ε, σχέδιο εφεδρικό και να γίνει και ο τριμερής διάλογο για να... Ε, γιατί ναι, όντω το κοινοβουλίο ψήφισε το Άμστερνταμ, αλλά υπάρχουν και κάποιες προποθέσει. Εκεί υπάρχουν προποθέσει προϋποθέσεις αυτές για κάποιο λόγο, δεν είναι τυχαίε. Να σας πω απλώς ότι και η Σουηδία είναι πολύ ωραία χώρα, εντάξει και θα μας ενδιέφερε και εμάς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, αλλά εντάξει δεν μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες, απλώς σας λέω ότι έχουμε και εμείς πάρα πολύ όμορφα μέρη στη δική μου τη χώρα. Και βέβαια παντού υπάρχουν ωραία μέρη, βορράς, νότος, ανατολή, δύση. Ο κύριος Βάλλη τώρα, ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Όσον αφορά την ε, υγιή δημοσιονομική διαχείριση, Ξέρετε ότι και στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής αλλά και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού δεν καταφέραμε να δούμε τις λεπτομέρειες της Ολλανδικής πρότασης διότι εκ των, προ... υστέρων μόνο μας δόθηκαν κάποια στοιχεία για το κόστος της έδρας στο Άμστερνταμ. Μας δόθηκαν κάποια στοιχεία από την ήδη φυστάμενη υπηρεσία στο Λονδίνο αλλά δυστυχώς δεν μας δόθηκαν καθόλου στοιχεία όσον αφορά την πρόταση της ε, Ολλανδίας. Μια πρόταση που ήταν τελικά πάρα πολύ αδιαφανής και που τελικά φαίνεται ότι θα κοστίσει πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα εκατομμύρια ευρώ σε τήσια βάση, χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αναλάβει και το Κοινοβούλιο της ευθύνη όσον αφορά την χρηματοοικονομική διάσταση της όλης υπόθεσης. Τώρα, πέρα από το κόστος αυτό, θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν τελικά η Ολλανδία θα καταφέρει να αποφύγει το επιπλέον αυτό κόστος το οποίο μας παρουσίασε. Έγινε μια αρχική πρόταση από την Ολλανδία που φαινόταν πολύ πιο οικονομική και εν συνεχεία οι κάτω χώρε υπέβαλαν μια άλλη πρόταση πολύ πιο δαπανηρή. Μα λέει αυτή τη στιγμή ότι θα οικοδομηθεί ένα νέο κτίριο, το οποίο δεν υπάρχει προφανώ ακόμα. Ενδεχομένω το τελικό κόστο θα είναι πολύ υψηλότερο από το πρώτο αυτό αρχικό κόστος το οποίο παρουσίασε στη δεύτερη πρότασή της η Ολλανδία. Νομίζω τα στοιχεία αυτά είναι ουσιαστική σημασία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σάλα, τώρα πάλι έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα να σας ξαναευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε. Με έχει συγκλονίσει η συζήτηση αυτή. Θα επιστρέψω στο Μιλάνο με ακόμα μεγαλύτερη την πεποίθηση ότι είμαι δυσαρεστημένος με τα όσα συνέβησαν. Μιλώ εξ ονόματος μιας από τις μεγαλύτερες ε, ευρωπαϊκές πόλεις και μια από τις πιο φιλοευρωπαϊκές πόλεις ε, αποδεικνύεται από τα γεγονότα, όχι στα λόγια. 15 μέρες ε, μετά από την εκλογή μου ως δημαρχού πριν δύο χρόνια πήγα στο Λονδίνο, διότι στην αίμα είδα ότι υπήρχε μια τεράστια ευκαιρία για την πόλη μου. Ζήτησα να επισκεφθώ κάθε γωνία του κτηρίου και από εκεί κινηθήκαμε. μα ζητήθηκε να συντάξουμε ένα φάκελο ολοκληρωμένο καλοφτιαγμένο, πλήρη και σήμερα το να μου λέει ο κύριος Κλάους ότι η Κομισιόν δεν κάνει συστάσεις δηλαδή ο φάκελος, η ποιότητα των φακέλων δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία και η ερώτησή μου είναι οι κυβερνήσεις όταν ψήφισαν γνώριζαν τους φακέλους γιατί μας ζητήσατε να συντάξουμε τόσο πλήρη φάκελο επενδύοντας δέσμευση πόρους, ενέργεια Εγώ ε, ε, έκανα άσχημη εντύπωση στους ε, πολίτες μου. Πήγα στους πολίτες μου και τους είπα πόσο σημαντικό ήταν να φέρουμε την αίμα στην πόλη μας και από τα όσα ακούω σήμερα ο φάκελος τελικά δεν έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Πόσο μάλλον που άλλαξαν και οι προποθέσεις. Εγώ λοιπόν ε, εκφράζω για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά μου. Ίσως να ακούσουμε και κάποιο σχόλια από την Κομισιόν, γιατί την ακούω, να, τη βλέπω να γνέφει το κεφάλι, να σχολιάζει κρυφά, να χαμογελά. Απαράδεκτη συμπεριφορά για Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω να πω ότι είμαστε φιλοευρωπαϊκή πόλη, στηρούμε τους κανόνες, τις αποφάσεις, αλλά είμαι απόλυτα απογοητευμένος από αυτά που άκουσα σήμερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, λείπαμε πάρα πολύ, αξιότιμε κύριε αλλά πρέπει να κλείσουμε τώρα το θέμα. Να επαναλάβω ότι στις 28 Μαρτίου φέτος ο δικός μας πρόεδρος ο Αντώνιο Ταγιάννη έστειλε μια επιστολή στο Συμβουλίο και στην Επιτροπή όπου επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο ο παρονθεσμός καταδικάζει απόλυτα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου δεν είμαστε καθόλου υπέρ. Θεωρούμε ότι δεν υπήρξε επαρκή δημοκρατική εξέταση τη διαδικασία αυτή, αυτής. Κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ ξανά. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε για αυτή την πολύ δυστυχή περίσταση. Θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Εγώ θα φροντίσω να πάει στον εισηγητή ε, κύριο Λαβία στις ε, Επιτροπές ΕΜΒ και ΑΦΚΟ για περαιτέρω εξέταση. Θα τους αναφέρουμε τα όσα ακούσαμε εδώ και επίσης θα ε, ενημερωνόμαστε διαρκώς για το τι συμβαίνει κατά την διάρκεια των τριμερών διαλόγων και επίσης θα μεριμνήσουμε ώστε όλοι να κατανοήσουν ότι η έλλειψη δημοκρατικής, ε, δημοκρατικού ελέγχου ε, επισημάνθηκε από εσάς όπως και από όλους, από όλες τις πολιτικές ομάδες. Κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Στο ψήφισμα της 15ης Μαρτίου το Κοινοβούλιο, ζήτησε να ενημερώνεται κάθε τρίμηνο για την κατάσταση του κτηρίου στο Άμστερνταμ και της κατασκευής του και των προσαρμογών κτλ. Ε, Εκεί θα θέλαμε να βλέπαμε περισσότερα, καλύτερη ενημέρωση. Αυτές οι εκθέσεις πρόοδου από την Επιτροπή θα πηγαίνουν στην ΕΜΒΗ και στον εισηγητή και θα κοινοποιούνται και στη δική μου Επιτροπή. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να αναλύει την υλοποίηση της κοινή δήλωση του 2012. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Εμείς θα πραγματοποιούμε ακόμη πιο συχνούς διαλογούς με τον εισηγητή και θα ακολουθήσουμε την νομοθετική διαδικασία για όλα αυτά και θεωρώ ότι η επίσκεψή σας εδώ σήμερα και η παρεμβάση σας ήταν κάτι πολύ επικαιρό και πολύ χρήσιμο όχι μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και ως υπενθύμηση προς το Συμβούλιο ότι αυτή η διαδικασία τύπου λαχιοφόρο αγοράς ε, είναι θλιβερή. Ε, πολλές αξίες ε, υπονομεύτηκαν με αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε εδώ. Πάρτε μαζί σας τον ήλιο των Βρυξελών και στο Μιλάνο επιστρέφοντας και μην διστάσετε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας για οτιδήποτε χρειαστεί. Είναι 12.30, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ.